Colleagues, we are starting. Να συνεχίσουμε συνάδελφοι. Φαίνεται ότι η Δημοσιονομική Επιτροπή είναι σε ένα πνεύμα συνεργασία. Ε, ξεκινήσαμε με μια κοινή συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ, ήταν το πρώτο σημείο τη ημερησία διάταξη, και το τελευταίο σημείο έχουμε κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και με την Επιτροπή Ανάπτυξη. Και συμπρόεδρο θα είναι ο κ. Στομπέ και θα συζητήσουμε το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Νομίζω ότι ε, είναι ε, πολύ σημαντικό να κάνουμε μία αξιολόγηση του νέου εργαλείου που συστήθηκε πριν δύο χρόνια και είναι κατάλληλη χρονική στιγμή πριν να πάρει την τελική του μορφή εν ώψη του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. Δεν ε, θα μακρηγορήσω λοιπόν, γιατί και πάλι δεν έχουμε πολύ χρόνο. 35 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. 10 λεπτά θα μας δώσουν παραπάνω διερμηνείς. Και θα δώσω κατευθείαν ε, το λόγο στον κύριο Τεμπέ για την εισαγωγή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Είναι εξαιρετική συνεργασία μεταξύ τριών διαφορετικών επιτροπών. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για να κερδίσουμε χρόνο. Για εμά η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αηφόρο ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους αναπτυξιακούς ε, στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη. Πρέπει από τα δις να πάμε στα τρεις, όπως θα γνωρίζετε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με, τη, με τους πόρους του ιδιωτικού τομέα. Το EFSD και ο διάδοχός του στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κοινοβούλιο έχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αυτού και έχει και νομοπαρασκευαστικό έργο και έτσι θα εμπλακεί στενά με αυτό το εγχείρημα. Δεν ήταν εύκολο, εύκολη η δημιουργία αυτού του Ταμείου για την αηφόρο ανάπτυξη. Ε, τα πράγματα δεν κινήθηκαν τόσο γρήγορα όσο θέλαμε στην αρχή. Χρειαζόμαστε λεπτομερείς πληροφορίες για το πόσες εγγύησεις έχουν κατοχυρωθεί, έχουν υπογραφεί, με ποιους εταίρους, με ποιους στόχους και πόσα ποσά κινητοποιούνται. Θα θέλαμε επίσης περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση αξιολόγησης του ταμείου αυτού την οποία έκθεση περιμέναμε στα τέλη του 2019 με βάση το άρθρο 17 του κανονισμού. Αυτή η έκθεση δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του Ταμείου αυτού, είναι καλό το γεγονός ότι γίνεται συζήτηση σήμερα, αυτή την περίοδο, για την τρέχουσα κατάσταση. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε και τη μελλοντική μας πορεία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, πιστεύω ότι Πρώτα πρέπει να προβούμε στην αξιολόγηση και μετά στη διαμόρφωση της νέας δομής αυτού του σχετικά νέου χρηματοδοτικού και χρηματοοικονομικού εργαλείου. Οφείλω να πω όμως ότι είμαστε κατά τη απογοητευμένοι για την κατάσταση. Διότι στις 21 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τη στρατηγική του. Ήταν η μέρα που συνεδρίασε και η δική μας Επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει καλύτερο συντονισμός αυτών των ε, ε, δύο οργάνων για να μπορούν τα μέλη μας που είναι παρόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο να μην χρειάζεται να είναι εδώ για λόγους επιτροπής αλλά να μπορούν να παρίστανται. Επίσης τα προπαρασκευαστικά έγγραφα, έγγραφα ε, καλό θα είναι να υπάρχουν ε, από πριν και να μην ε, δημοσιεύονται μετά τις συνεδρίες και τη σύσκεψη του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ταμείου αυτού. Έχουμε την κυρία Μαριέτα Γιάκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Προπολογισμών και Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Από τρει επιτροπέ είστε παρόντε σήμερα και είναι πολύ μεγάλη τιμή που μπορώ να σα αναφέρω την πρόοδο σε σχέση με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αϊφόρο Ανάπτυξη και να σα μιλήσω για τι εγγυήσει που έχουν υπογραφεί και τις συμφωνίες με βάση το εφιστάμενο επενδυτικό σχέδιο και πρόγραμμα. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι χάρη στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο υιοθετήσαμε το σχετικό κανονισμό το 2017 σε ένα χρονικό διάστημα ρεκόρ, εξαιρετικά βραχή και βλέπω μέλη του Κοινοβουλίου παρόντα, τα οποία διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές και στον τριμερή διάλογο τότε, ο οποίος μας επέτρεψε να προχωρήσουμε εξαιρετικά γρήγορα, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά θετικό σημαντικό. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα μέρη ε, τη έκθεση αξιολόγηση τα οποία θα σα διαφυβάσουμε. Πιστεύω ότι σα το έχω ήδη πει αυτό γιατί δείχνουμε τι επιτυχίε αυτού του ταμείου επίσης δεν είναι καθόλου ασήμαντες στο βραχή χρονικό διάστημα της ύπαρξής του. Και έχω ετοιμάσει και κάποιε διαφάνειε, οι οποίε υποστηρικτικά θα λειτουργήσουν. Τέσσερι ήταν οι συσκέψει του ε, Στρατηγικού Συμβουλίου. Πάντοτε και στι τέσσερι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν προσκεκλημένο. Λυπούμαστε βαθύτατα διότι ε, στις 21 Ιανουαρίου στην τελευταία σύσκεψη εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου δεν μπόρεσε να παραστεί. Εμείς ορίσαμε αυτή την ημερομηνία γιατί είχαμε τις τέσσερις υπογραφές την ίδια ημέρα και στη συνέχεια εκ των υστέρων μάθαμε ότι η Επιτροπή ΔΕΒΕ δεν μπορούσε να αναβάλει τις εργασίες της για άλλη μέρα προκειμένου εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου να έρθει και σε εμά. Σας υποσχόμαστε ότι θα συντονίσουμε καλύτερα τα πράγματα την επόμενη φορά. Θα ήθελα να μπει η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ και να πω ότι το Ταμείο ξεκίνησε με μια, ε, έκανε μια λαμπρή αρχή θα έλεγα και έχουμε 7 ε, συμφωνίες εγγυήσεων, εγγυητικές συμφωνίες και έχουμε ε, με έναν πυλώνα πολύ βασικό με αρχή το 2018 το Επιχειρησιακό Συμβούλιο ενέκρινε 28 προτάσεις για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα με βάση 5 εγγυητικά παράθυρα. Ίσως σας ε, εμπλέκουν λίγο οι όροι αυτοί, γιατί βλέπετε από τη μία το εξή νούμερο, 1,57 δις και θα θυμάστε από τον κανονισμό για το Ταμείο για την Αϊφόρο Ανάπτυξη προβλέπεται εγγύηση για 1,5 δις. Υπάρχει μια μικρή απόκληση λοιπόν και με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι έχουμε δεχθεί επιπρόσθετες συνεισφορές. 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ίδρυμα Gates, 10 εκατομμύρια ευρώ από τη Δανία και επιπρόσθετη συνεισφορά από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γερμανία και την Εσθονία, τα οποία ε, ποσά έχουν αφιερωθεί και τεθεί κατά μέρος για ψηφιακά ε, project και προγράμματα. Και βλέπετε ότι με την κατανομή αλλά με τις, και με τη μόχλευση θα φτάσουμε στα 7,5 δις, θα δημιουργηθούν 4 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, θα απαλληλθεί μεταναστευτική πίεση γυναικών και παιδιών, θα μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα και με χαρά σας αναφέρω ότι η γεωγραφική κατανομή των πόρων ε, συμφωνεί με τους νομοθέτες, με εσάς. Δύο τρίτα για την υποσαχάρια Αφρική και ένα τρίτο για τις γειτονικές όμορες περιοχές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασική τομή, αϊφόρος, ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερος τομέας, γυναίκες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε βρει και επιπρόσθετα κονδύλια άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ για τεχνική βοήθεια. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να στήσουμε σωστά το τρίτο πυλώνα, να έχουμε ένα στέρεο νομοθετικό περιβάλλον ε, το οποίο είναι απαραίτητο για να έχουμε ε, βιώσιμες επενδύσεις και ε, αφιερώσαμε 700 εκατομμύρια σε αυτό το κανονιστικό σκέλος, το κομμάτι που έχει να κάνει με τις διατάξεις και το νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο. Μπορώ να σας μιλήσω τώρα για τις αποφάσεις του Στρατηγικού Συμβουλίου το οποίο ενέκρινε τις επενδυτικές περιοχές, τα οποία ε, αναφέρουμε ως ενεργειακά, ενεργει, επενδυτικά παράθυρα. Έχουμε την εγγύηση, ε, το τζίτα, την ομάδα για την τεχνική αξιολόγηση των εγγυήσεων, αυτό είναι το τζίτα, και υπογράψαμε αυτές τις 7 εγγυητικές συμφωνίες. Ξεκινήσαμε στα τέλη του 2018 στη Βιέννη με τον Αζίρα, μια πολύ σημαντική εγκυητική συμφωνία, η οποία δημιουργήθηκε ώστε να βοηθήσει τους Σύρους πρόσφυγες στην Ιορδανία. Μιλούμε για 75 εκατομμύρια, εγγυήσεις ύψους 75 εκατομμυρίων. Μιλούμε για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο βοηθά στην αποκοινού ανάληψη του κινδύνου και έχουμε και μια δεύτερη φορά συμφωνιών εγγυητικών που υπογράφησαν για περαιτέρω βοήθεια για πρόσφυγες στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που τους βοηθούν για το κατάλημα και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για αυτούς. Στη συνέχεια, στο Γιωχάνεσμπουργκ, το Νοέμβριο του 2019, υπογράψαμε το Αρχιπέλαγος, μια εγγυητική συμφωνία, αλλά και το Capital Venture με το FMO. Το αρχιπέλαγος με το CDP έχει ύψους 30 εκατομμύρια και το ε, ε, Common Venture έχει ύψος κονδυλίων 42 εκατομμύρια. Έχουμε τέσσερις υπογραφές οι οποίες έπεσαν ε, στις 21 Ιανουαρίου φέτος. Συνέβησαν ταυτόχρονα δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντική συμφωνία την Ρεζίντα ύψους 100 εκατομμυρίων και Υπογράψαμε μια συμφωνία ε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, την EBRD. Όλα αυτά μαζί λοιπόν δείχνουν ότι έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει 357 εκατομμύρια από τις ε, διαθέσιμες εγγυήσεις, περίπου το 1 τέταρτο ε, των εγγυήσεων για τις οποίες γίνεται λόγος. Θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια τώρα μάλλον στην προηγούμενη πήγατε δύο πιο μετά, ενώ εγώ θα ήθελα μία την επόμενη μόνο. Πρέπει να πάτε μία πίσω. Να σας δείξω ότι είναι διαφοροποιημένη η χρηματοδοτική αρχιτεκτονική. Συνεργαζόμαστε με 10 διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πιστεύουμε ότι η συνεργασία με πολλούς εταίρους είναι αυτό το οποίο κομίζει ποιότητα στο εγχείρημά μας. Ε, σημειωτέων ότι 1,5 δις, εγγύησης ύψους 1,5 δις, ε, καλύφθηκαν τρεις φορές με τις προτάσεις που δεχθήκαμε. Δηλαδή ζητήθηκε τρεις φορές περισσότερο από τη δική μας πρόταση. Και ως προς τη μόχλευση, τελικά ε, μοχλεύουμε ε, ποσά εγγύσεων ύψους 17,5 δις στην υποσαχάρια Αφρική και στην εγγύς Ανατολή. Τώρα, θα με ρωτήσετε γιατί μόνο 7 σας απαντώ λέγοντα ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει τέτοιου είδους εγγυητικέ συμφωνίες με κάποιο εξωτερικό μέρος, τρίτο μέρος και υπάρχει και εμπορικό σκέλο στι συμφωνίε, το οποίο συντάξαμε με τη βοήθεια μιας πολύ καλής δικηγορικής εταιρείας δεν ήταν τόσο μεγάλη πρόκληση τα οριζόντια ζητήματα που χρειάστηκε να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ε, τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες μας, π.χ. την ε, πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο και το καθεξής. Τα επόμενα τώρα βήματα είναι τα εξής. Θα προσπαθήσουμε να υπογράψουμε 8 ακόμα τέτοιου είδους συμφωνίες μέχρι το καλοκαίρι και τις υπόλοιπες να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το Δεκέμβριο. Διότι, όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός προβλέπει ότι όλες οι συμφωνίες πρέπει να έχουν συναυθεί και υπογραφεί μέχρι τα τέλη του 2020. Τώρα, όλες οι προτάσεις που δεν έχουν ακόμα ε, ξεκινήσει είναι σε αμναμονή ε, θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις μέχρι την 28 Φεβρουαρίου. Και θα ήθελα να μιλήσω για το EFSD blending με το EIP, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια για να βρούμε τα χρήματα σε γεωγραφικά προγράμματα, για να τα βάλουμε σε αυτό το blending, σε αυτό το μείγμα. Ε, βάλαμε 3,1 δις που μποχλεύονται και ανέρχεται το ποσό της μόχλευσης στα 30 δις για 154 project που θα χρηματοδοτηθούν ε, στον τομέα των μεταφορών της ενέργειας, της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και της γεωργίας στην υποσαχάρια Αφρική 78 τέτοιου είδους έργα και στην γειτονιά, στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 76 ε, προγράμματα περίπου και είμαστε πολύ απασχολημένοι με τις ε, δραστηριότητες επικοινωνίας, επίσκεψης, επαφής με το κόσμο. Δεν θέλουμε να είμαστε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολλές αντιπροσωπείες και αποστολές. Το 2019 είδατε, βλέπετε πόσες ε, ε, εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος οργανώσαμε στις διάφορες αυτές χώρες, Καμερούν, Αγκόλα, την Ισία, Σενεγάλη, Σχέρα Λεόνε. Το 2020 προγραμματίζουμε στην Ουκάντα, στην Μπουρκίνα Φάσο, μεταξύ μεταξύ άλλων στη Μαδαγασκάρη και σας καλώ να έρθετε να παραστείτε σε, αυτές τα, σε αυτά τα business events στις χώρες αυτές για να δείτε πώς εφαρμόζουμε το ε, σχέδιό μας για εξωτερικές επενδύσεις. Επιτρέψτε μου τώρα να πω δύο λόγια για την αξιολόγηση. Ζητώ συγγνώμη για την ε, ελαφρά καθυστέρηση που παρουσιάζει η δημοσίευση των ανακοινώσεων ε, και των αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση. Ε, αργήσαμε γιατί θελήσαμε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό κείμενο. Μπορώ όμως ήδη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σχετικές συστάσεις και συμπεράσματα της έκθεσης που σας αφορούν. Λέει λοιπόν η έκθεση στην οποία καταλήξαμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αεφορό Ανάπτυξη ενδιαφέρει άμεσα σε σχέση με τα προαπαιτούμενα που προβλέπονται στο νέο μοντέλο παγκόσμιας ε, ε, ε, χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει μια νέα γενιά δωρητών. Τώρα για την αποτελεσματικότητα και την αθρηστικότητα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αϊφόρο Ανάπτυξη συγκεντρώνει σημαντικά κονδύλια για τη μόχλευση με δίκτυ 10 τα στοιχεία δείχνουν ότι διευκολύνεται έτσι η διοίκηση με διαφάνεια. Ε, περισσότερη διαφάνεια στο management δηλαδή. Είναι πάρα πολλά τα συμπεράσματα τα οποία είναι θετικά. Ε, σας τα παραθέτω και σας τα διαβάσω ε, εντάχει. Το Ταμείο αυτό ενθαρρύνει μεγαλύτερο συντονισμό και ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των προσπαθειών Πρέπει να έχουμε το μοντέλο της ανοιχτής πρόσβασης, μεγαλύτερη μίξη μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η αξιοπιστία μας. Αυτά προς το παρόν. Με χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είναι καλό να έχουμε θετική αξιολόγηση εξωτερικών δημοσιονομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τον, τις καθοριστικές διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις στις 20 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τώρα να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Βαρδία Σαμπάλ. Από τις τρεις ε, είναι παρούσα και νομίζω ότι όλοι οι φάκελοι είναι δικοί σας, είστε αρμόδια για όλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι αυτά που έχουν τελικά συσσωρευτεί από την προηγούμενη θητεία και κάποιο τελικά πρέπει να ασχολείται με όλα αυτά. Καταρχήν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι πληροφορίε και φυσικά και για τη δουλειά σα. Ε, είναι αλήθεια ότι διαπραγματευόμασταν αυτό το ταμείο και βλέπουμε τώρα το να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό είναι αρκετά θετικό και στην παρουσίασή σας είδα να αντικατοπτρίζονται λέξεις και ιδέες που επεξεργαστήκαμε εμείς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν ε, προγράμματα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, να επικεντρωνόμαστε στις γυναίκες, τους νέους, στην Ήπεθρο και ξέρετε φυσικά ότι αυτό το κοινοβούλιο πάντοτε ε, τα υπεράσπιζε αυτά και γι' αυτό το τονίσατε κι εσείς στην παρουσίασή σας. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι εργαζόμαστε στους τομείς ε, που είπαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο μέσο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είχα κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τις ημερομηνίε και με την τεκμηρίωση που πρέπει να λάβουμε. Εκ των προτέρων όμως το είπε εδώ ο Πρόεδρος και νομίζω το σημείωσε η Κομισιόν. Έτσι λοιπόν δεν θα αναφερθώ σε αυτά, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, είναι αλήθεια ότι καθυστερήσατε αρκετά για να υπογράψετε τις πρώτες συμβάσεις και είναι λογικό όταν ε, τίθεται σε λειτουργία ένα νέο μέσο όμως, όπως σχολιάσατε, εργαζόμαστε για το μελλοντικό μέσο, ακόμη δεν έχουμε διαθέσιμη αυτή την αξιολόγηση, αλλά είναι αλήθεια ότι θα θέλαμε να βελτιώσουμε το επόμενο μέσο όπως μπορούμε. Και θα ήθελα λοιπόν να, πού, να ρωτήσω πού είχατε δυσκολίες και γιατί άργησαν να το συνυπογραφούν αυτές οι πρώτες συμβάσεις εγγύησης. Τώρα, σε σχέση με το προσωπικό που, θα, που έπρεπε η Κομισιόν να θέσει στη διάθεση αυτού του μέσου και για το μελλοντικό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ΣΥΝ. Ε, σίγουρα θα χρειαστούν ε, ε, περισσότεροι δικοί για αυτή τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι βήματα κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως έχοντας κατά νου ότι η πρόταση που υπάρχει επιτάπητος θέλει να κόψει πολύ και ε, το προσωπικό της διοίκησης. Εμείς ε, θα θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό γιατί τελικά τα βαραίνουμε τα προγράμματα. Τρίτον, είναι αλήθεια ότι συζητήσαμε πολύ και αναφερθήκατε και στην παρουσίασή σας στο θέμα της μόχλευσης των προγραμμάτων. Όμως ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Σημαντική είναι η μόχλευση και γι' αυτό έχουμε τέτοια χρηματοοικονομικά μέσα. Όμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε σημαντικά προγράμματα που έχουν μικρότερη μόχλευση αλλά που έχουν ε, πιο θετικές κοινωνικές επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν ε, θα θέλαμε να μας εφησυχάσετε κάπως ε, στο θέμα αυτό και να μας πείτε ότι λαμβάνετε υπόψη όχι μόνο το οικονομικό σκέλος αλλά και το κοινωνικό σκέλος. Και καθώς αξιολογείτε τα διάφορα προγράμματα και απορρίπτετε κάποια προγράμματα χρηματοδότησης, ε, θα ήθελα να τα λάβετε αυτά υπόψη. Και νομίζω θα σταματήσω εδώ γιατί ήθελα πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ φυσικά προσυπογράφω όλα σε είπε η που ήταν μία από τους πρωταγωνιστές της δημιουργίας αυτού του ταμείου. Τώρα για το χρόνο και τον τρόπο ε, πράγματι ε, θέλουμε να γνωρίσουμε πολύ περισσότερα γιατί και από την Επιτροπή ΔΕΒ είχαμε επενδύσει πάρα πολύ στην πρόταση αυτή. Και μάλιστα είχαμε φανταστεί ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και μια διαφορετική οργάνωση από ό,τι συμβαίνει στα παραδοσιακά εργαλεία ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα ε, εξαίρετο μέσο. Θα ήθελα να καταλάβω όμως λίγο περισσότερα γιατί ε, σίγουρα συμφωνούμε επί των προγραμματών και των θεμάτων, ε, ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, γυναίκες, νέοι, όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά. Όμως, για να καταλάβουμε πώς θα δημιουργήσουμε μία αηφόρο ανάπτυξη και όχι εφήμερες εμπειρίες, δηλαδή όταν τελειώνει η εξωτερική δράση, μας να μην μένει το κενό και να μην το αισθάνεται έτσι και τοπικές κοινότητες. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εργαστήκατε έτσι ώστε να υπάρχει και ένα στοιχείο βιωσιμότητας, αυτονομίας και διάρκειας στο χρόνο των προγραμμάτων και να μας πείτε πώς ακριβώς εκπαιδεύετε τους τοπικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή τους μικρούς επιχειρηματίες. Ε, προκειμένου οι ίδιοι να έχουν την ικανότητα στη συνέχεια να δώσουν μια συνέχεια στα προγράμματα. Ποιο ρόλο λοιπόν παίζει η κατάρτιση του τοπικού προσωπικού των ανθρώπων που επιτόπου μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτόν τον προγραμματισμό των έργων. Ναι, έχετε δίκιο. Το Ταμείο για την Αϊφόρα Ανάπτυξη θα πρέπει να υποστηρίζει αϊφόρα προγράμματα. Τώρα η Κομισιόν για να μας απαντήσει. Thank um, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και ασφαλώς και εκτιμούμε το θέμα της ερωτήσης που θέσατε. Συμμεριζόμαστε και τις ανησυχίες σας για το κοινωνικό σκέλος το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο τον παράγοντα αμόχλευσης. Γι' αυτό λοιπόν ε, ρυθμιζόμαστε ανά κλάδο και αναχώρα, αλλά ξέρετε τι γίνεται και με την τιμολόγηση. Σε ό,τι αφορά τα λύσεις, για παράδειγμα, όταν κινηθούμε στους τομείς και στους κλάδους που χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παρέμβαση, μπορούμε να προβούμε και σε νομοθεσία. Ναι, σε ρύθμιση, Να πω ότι ω τώρα, σε όλα τα παρατήματα όλων των συμφωνιών, η Οι ρήτρε αυτές ακολούθησαν ε, τις ε, σχετικέ για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και θέσαμε λοιπόν τις προτεραιότητες μας ανά τομέα και αυτό σε, σε ό,τι αφορά και τις βιώσιμες πόλεις, τη βιώσιμη ενέργεια, τη βιώσιμη συνδεσιμότητα γιατί πρόεδρε και αγαπητοί βουλευτές αυτό είναι η αηφορία το συζητάμε αυτό και με τα άλλα δημοσιονομικά όργανα. Θα πρέπει να υπάρχουν βιώσιμε επενδύσει προκειμένου να ξεπεραστούν τα ζητήματα. Από πλευρά μα αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει τοπική παρουσία, να έχουμε ε, με... στρατεύματα επιτόπου. Προκειμένου να υπάρχει μια, ένα, μια μόνιμος, μόνιμος αντίκτυπος. Και εξετάζουμε τη δυνατότητα να κοιτάξουμε για το EFSD+, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+, να κοιτάξουμε και τη Λατινική Αμερική και την Ασία, να δούμε και άλλε δυνατότητε. τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει να δούμε και το ψηφιακό σκέλο σε ό,τι αφορά την Πράσινη Συμφωνία, σε ό,τι αφορά τμήμα των βαθύτερων αιτιών ε, για την μετανάστευση. Χρειάζεται λοιπόν ε, ίδια μόχλευση και η κάθε μόχλευση να έχει το ίδιο αντίκτυπο. Θα επιδείξουμε όμως ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μόχλευσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το 50%. Τον όρο 50% θα πρέπει να υπάρξει μόχλευση σε κάθε κλάδο και να υπάρχει αντίστοιχο επίπεδο παντού. Ήθελα να το αναφέρω αυτό. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να καθορίσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μέλλοντος. Α, ξέχασα να αναφέρω ότι χρησιμοποιούμε και την τεχνική αρρωγή ασφαλώ και το κλάδο των επιχειρήσεων για να υπάρχει πραγματικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος της EIP το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σίγουρα ο όρος που χρησιμοποιούμε περισσότερο σήμερα το απόγευμα είναι ο όρος βιώσιμος και η μόχλευση είναι ο δεύτερος όρος. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τομπέ για καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Να πω ότι σίγουρα οι μελλοντικοί μήνες θα είναι πολύ ενδιαφέροντες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τις ε, ευκαιρίες ε, που προσφέρονται. Αν ε, μπορέσουμε επιτυχώς να συντονίσουμε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα με εμπειρογνωμοσύνη, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε κανονιστικό πλαίσιο και διαφανά θεσμικά όργανα και μπορούμε να, επενδύ, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους και φυσικά καλό είναι να έχουμε την αξιολόγηση και μπορούμε να τη λάβουμε απόψη για τη μελλοντική δουλειά μας. Νομίζω ότι εδώ όμως προσφέρονται κάποιες ευκαιρίες και ελπίζω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή σύμφωνα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας και φυσικά θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με πάρα πολύ ενδιαφέρον.